αυτή τώρα η ψηφοφορία σήμερα με απλοποιημένη διαδικασία για την έκθεση τη κυρία Ματιέ για το Μουσουλμικό έλεγχο των κονδυλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη τη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ναι, καθίστε παρακαλώ στι θέσει σα. Ψήφισαν όλοι. Πέραση τη ψηφοφορίας. Ορίστε, κυρία μου, σας ευχαριστώ. 550 υπέρ, 5 κατά, οπότε εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην κυρία Ματιέ. Έκθεση Ριέρα Ματζουρέλ για την εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Έχουμε το σχέδιο ψηφίσματος. Έχουμε τροπολογία 3, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι, ψηφίσατε αγαπητές συνάδελφοι, πέρας τη ψηφοφορίας. 537 υπέρ, 22 κατά, γίνεται δεκτή η τροπολογία. Αυτή ήταν όλη η ψηφοφορία. Συγχαρητήρια στην κυρία Ριέρα Μαντουρέλ. Περνάμε στην ψηφοφορία για τα γεγονότα στην Γάζα. Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ. Σούλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε εσείς και οι συνάδελφοι δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα μία για το ψήφισμα το οποίο βρίσκεται μπροστά μας και μετά μία προσωπική παρατήρηση που απευθύνεται στους συναδέλφους. Πρώτα απ' όλα για το ψήφισμα. Η ομάδα μου, κυρίες και κύριοι, χτες το βράδυ συζήτησε έντονα και με πολύ πάθος και πολύ σοβαρά αυτό το ψήφισμα. Πριν ψηφίσουμε, είμαι σίγουρο σήμερα πως όλοι είμαστε εντυπωσιασμένοι από αυτά τα οποία μόλις ανέφερε ο Φράνσις Βούρτς. Δηλαδή, εάν πλέον ούτε και οι διεθνείς οργανισμοί δεν γίνονται σεβαστοί και δεν είναι ασφαλείς, έχουμε φτάσει στο σημείο στο οποίο πρέπει να απευθύνουμε έκκληση στο Ισραήλ να σεβαστεί τους διεθνείς οργανισμούς αλλιώς ε, δεν είναι δυνατό να εγγυηθούμε τις ε, ε, ανθρωπιστικές συνθήκες έχουμε μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου απ' την άλλη όμως αποφασίσαμε να στηρίξουμε αυτό το ψήφισμα γιατί μετά από μεγάλη συζήτηση χτες το βράδυ γιατί θεωρούμε πως είναι σωστό αυτή τη στιγμή να το εγκρίνουμε και γιατί το μήνυμα το οποίο εμείς και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στείλουμε ε, πρέπει να είναι το εξής ότι εάν φτάνουμε στο να μην γίνονται σεβαστά πλέον και να βομβαρδίζονται σχολεία και νηπιαγωγεία δεν μπορεί να μιλάμε για λύπη. Είναι κάτι που πρέπει να καταδικάσουμε. Το δεν βρίσκεται στο ψήφισμα, αλλά επειδή θεωρούμε πως αντικατοπτρίζουμε και τα συναισθήματα πολλών συναδέλφων και από άλλες ομάδες, πως πρέπει να αναφερθεί Και θα ήθελα να αφαιρθώ σε έναν ε, συνάδελφο ο οποίος έχει συνεισφέρει πάρα πολλά και στην παγκόσμια ειρήνη κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Πρόκειται για την τελευταία του Ολομέλεια, πρόκειται για τον συνάδελφο τον Μισελ Ροκάρ. Για εμάς σοσιαλιστές λοιπόν, αλλά και για όλους πιστεύω, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω προς τον ε, κύριο Ροκάρ δεν μπόρεσα να είμαι παρόν χτες στην ε, δεξίωση γιατί ήταν εδώ ο κύριος Τοπολάνεκ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας κύριε Ροκάρ, την φιλία μου και σας εύχομαι Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ελπίζω να σας ξαναβλέπουμε συχνά και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτά τα οποία έχετε προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ κύριε Μισελ So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Gala möchte eine mündliche zu... Θα ήθελε ένα συνάδελφο να κάνει μια προφορική τροπολογία στο σημείο 3. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σε συνεννόηση και με τις άλλες ομάδες θα ήθελα να προτείνω την εξή τροπολογία. Στα αγγλικά του replay να αντικατασταθεί το ειδική ευθύνη με τον σημαντικό ρόλο έτσι ώστε η πρόταση να έχει ως εξή. Κάτι το οποίο υπονοεί ένα σημαντικό ρόλο για την Αίγυπτο. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση οπότε ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ, σηκώστε το χέρι. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές. Αν βλέπω καλά με μία αποχή, εγκρίνεται λοιπόν. Ψηφίζουμε άρα την αιτιολογική σκέψη γάμα σε δύο ξεχωριστά τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Δέλτα. Όχι, γάμα. Το σωστό μου λέει πάντα ο συνάδελφος. Ναι, ναι, αλλά ε, μου λένε από κάτω και σοβαροί συνάδελφοι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πρώτο του γάμα, υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές, δεκτό. Μπορούμε να το εξετάσουμε έναρξη της ψηφοφορία Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Abgestimmt. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 353 υπέρ, 214 κατά. Γίνεται δεκτό. Ψηφίζουμε τώρα το κείμενο, το σύνολο του ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές με λίγες αποχές και καμία ψήφο κατά εγκρίνεται το κείμενο. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πληροφορήσω πως τώρα θα αναλάβω μια προσπάθεια ως πρόεδρος της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης να έχουμε ένα ανάλογο ψήφισμα και στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Διάσκεψη με αυτό το οποίο εγκρίναμε εδώ σήμερα. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα για το κέρας της Αφρικής. Υπάρχει μια πρόταση ψηφίσματος από έξι ομάδες. κυρία Γκόμες θέλει να καταθέσει μια προφορική τροπολογία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θέλω να προτείνω μια νέα παράγραφο πριν το ένα που θα λέει τα εξή. Σημειώνουμε ότι η φυστάμενη κατάσταση στις χώρες του κέρατος της Αφρικής δεν συμβαδίζει με τα βασικά στοιχεία της συνεργασίας που περιλαμβάνει το άρθρο 9 της Συμφωνίας Κοτονού. Πρόκειται για μια φράση που ήταν ήδη στην έκθεση που περιλάμβανε, που είχαν συντάξει τρεις συνάδελφοι που περισκέφθηκαν την περιοχή πρόσφατα. Ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ, ο κύριος Νασάουρ. Okay, the... Με μικρόφωνο, παρακαλώ. Η ομάδα του ΕΛΚ είναι κατά της προφορικής τροπολογίας. Ναι, ναι, σηκωθείτε, παρακαλώ. Ναι, είναι 40 συνάδελφοι. Οπότε ψηφίζουμε. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το σημείο 1, οπότε Περνάμε στην τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 7 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ. Ευχαριστώ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 3 υπέρ. Ευχαριστώ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε το συνολικό σχέδιο ψήφισματος με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. 570 υπέρ, 11 κατά, εγκρίνεται μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ όλους ε, όσου συνεργάστηκαν. ακολουθεί η ψηφοφορία για τι πέντε προτάσεις ψηφίσματο για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Έναντι της ε, Λευκορωσίας. Ψηφίζουμε πρώτα απ' όλα το σημείο 9, ο Μαρίνος Βίρτς μας, σημείο 9, θα ήθελα να κάνει μια προφορική τροπολογία. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Προτείνουμε την διαγραφή της τελευταίας παραγράφου, της, της τελευταίας φράσης στην παράγραφο 9 που αναφέρει «Καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να θέσουν τέρμα στην πρακτική τους να διεκδίδουν θεωρήσει εξόδου στους πολίτες της χώρας και ιδίω στα παιδιά και τους φοιτητέ. Θέλουμε να φύγει η πρόταση αυτή διότι το σύστημα θεωρήσεων εξόδου έχει ήδη καταργηθεί από τις αρχές της Λευκορωσίας. Ευχαριστώ. Οπότε προφορική τροπολογία στο σημείο 9 δεν υπάρχει αντίρρηση οπότε την ψηφίζουμε ποιο είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχέ Δεκτή. Τροπολογία 1 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Πρέπει να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 242 υπέρ, 340 κατά, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου ψηφίσματος, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 551 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ όλους όσους εργάστηκαν γι' αυτό. Ψηφίζουμε τώρα κοινή πρόταση ψηφίσματο έξι ομάδων που αντικαθιστά όλε τι προηγούμενε προτάσει για την Σερεμπρέντσα. Η κυρία Ντόρι Πακ θέλει να καταθέσει προφορική τροπολογία για το σημείο 3. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι υπερψήφισαν την αντικατάσταση του σημείου 3. Το σημείο 3 αφορά την αποστολή του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Θέλουμε να συμπληρώσουμε την εξής πρόταση στα αγγλικά. Επαναλαμβάνει Είπα αυτή τη σκοπιά πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εγκλήματα πολέμου στο ε, εσωτερικό επίπεδο. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση οπότε ψηφίζουμε το σημείο 3 όπως έχει. Α, όχι, ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία όλη την πρόταση ως έχει έναρξη της ε, ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 556 υπέρ, 9 κατά. Γίνεται δεκτό σας. Ευχαριστώ όλους. Περνάμε τώρα στις δηλώσεις. επεξηγήσεις ε, ψήφου. Πρώτα απ' όλα για την έκθεση Ριέρα Μαντουρέλ, συνάδελφος Χένεν.